λαϊκή δημοκρατία της ναι, Βορείου ναι. Και τώρα προχωράμε στην ε, ε, συνεδρίασή μας. Τα πρακτικά της ε, χθεσινής ολομέλειας είναι στη διάθεσή σας. Έχετε παρατηρήσεις, δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Εγκρίνονται.